Okay. Uh, good afternoon. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, λέει Πρόεδρος. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να καλωσορίσω εδώ τον κύριο Όλαφ Σόλτς, Πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ και Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών και Αντικαγκελάριο της Γερμανίας για τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε όσον αφορά τις προτεραιότητες του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα θα συζητήσουμε και για την κρίση της πανδημίας COVID-19. Κάτι το οποίο αποτελεί βέβαια μια υγειονομική κρίση, αλλά έχει και τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία μας και στην καθημερινότητά μας. Το βλέπουμε αυτό, το νιώθουμε και από το Μάρτιο όλες οι χώρες μέλη έχουν υιοθετήσει μέτρα για να στηρίξουν την εθνική τους οικονομία και για να διασφαλίσουν όσο γίνεται περισσότερο την ευημερία των νοικοκυριών και των πολιτών γενικότερα. Αυτή η προσπάθεια συνοδεύτηκε και από σημαντικέ πρωτοβουλίε που ανελήφθησαν αμέσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το πακέτο για την ανάκαμψη σίγουρα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προ αυτή την κατεύθυνση και σε αντίθεση με αυτό που έγινε το 2008 όταν ξέσπασε τότε η κρίση, αυτή τη φορά ανταποκριθήκαμε αμέσως και ήταν σαφές ότι το πακέτο αυτό θα έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω από τη συσσόρευση απλώς και την πρόσθεση των εθνικών προσπαθειών. Όλα αυτά τα μέτρα σίγουρα διευκόλυναν την δράση των εθνικών κυβερνήσεων και έτσι δεν κατέρευσε η οικονομία. Παρόλα αυτά όμως, όπως βλέπουμε από τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα αυτά θα οδηγήσουν σε μία άνηση βέβαια, αύξηση του χρέους των χωρών μελών όσον αφορά τη σχέση του με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Ακριβώς αυτές οι διαφορές οφείλονται και με, από το, στο πώς χτύπησε η πανδημία την κάθε χώρα, αλλά και το πώς μπόρεσε να αντισταθεί κάθε χώρα. Οι χώρες μέλη, λοιπόν, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτήν την οικονομική κρίση και τις συνέπειες του COVID-19 της πανδημίας με τα ίδια μέσα και με την ίδια δύναμη. Κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μεγάλη διαφοροποίηση μέσα στην Ευρωζώνη, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε ήδη, ότι θα υπάρξουν αρνητικές ε, επιπτώσεις, αρνητικός αντίκτυπος με πιέσεις. Το πακέτο λοιπόν για την ανάκαμψη προσπαθεί ακριβώς να αντιμετωπίσει αυτές τις ε, προκλήσεις. Ήταν φιλόδοξη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσον αφορά το συνολικό πακέτο αλλά και όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις που προτάθηκαν. Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο του Ιουλίου και χαιρόμαστε βέβαια ήδη για τα αποτελέσματα, παρόλα αυτά μας απογοήτευσε σε έναν βαθμό γιατί προτείνει περικοπές στα κονδύλια και μάλιστα κατάργηση κάποιων προγραμμάτων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αποτελούν κλειδί για να μπορέσουμε να στηρίξουμε με εναρμονισμένο τρόπο την μάχη που δίνουν οι χώρες μέλη. Είναι σημαντικό λοιπόν να είναι ξεκάθαρο για όλους μας ποιοι είναι οι στόχοι του σχεδίου ανάκαμψης, που είναι να καλύψουν τα κενά τα οποία προκύπτουν εξαιτία της πανδημίας COVID και συγχρόνως να αντιμετωπίσουν κάποιες από τις διαφορετικές αδυναμίες των οικονομιών των χωρών μελών έτσι ώστε να υπάρξει σύγκληση και να ενθαρρύνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το πακέτο ανάκαμψης πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία, είναι μια ευκαιρία για να ξαναχτίσουμε τις οικονομίες μας σε πιο γερά θεμέλια, με ανάπτυξη που θα κρατήσει χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη μας βέβαια την πράσινη διάσταση, την βιωσιμότητα και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να διατηρήσει και να ενισχύσει την θέση της που είναι στην πρώτη γραμμή. Να ξέρετε ότι εμείς θα βοηθήσουμε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σόλτς, λοιπόν, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω τη διαδικασία για την ανταλλαγή αυτή απόψε. Πρώτον, λοιπόν, θα έχουμε εισαγωγικέ παρατηρήσεις από τον κύριο Σόλτ. το πολύ 15 λεπτά. Και στη συνέχεια ε, θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. 10 ερωτήσεις και απαντήσεις συνολικά, 5 λεπτά κάθε μία, 2 λεπτά δηλαδή για την ερώτηση και 3 λεπτά για την κάθε απάντηση. Και σας παρακαλώ όλους να τηρείτε το χρόνο σα. Είναι δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, εξ αποστάσεως, όπως βρίσκομαι εγώ, να παρεμβαίνω και να σας θυμίζω ότι έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας. Στον πρώτο γύρο η κάθε πολιτική ομάδα θα έχει μία ερώτηση και μία απάντηση ε, και μετά θα εφαρμόσουμε το σύστημα DONT, ανάλογα δηλαδή με το βάρος κάθε πολιτικής ομάδας. Και αν έχουμε χρόνο, μετά θα χρησιμοποιήσουμε και τη διαδικασία Catch the Eye. Συνεπώς, επίσης θυμίζω ότι έχουμε διερμηνία Φροντίστε να μιλάτε καθαρά, παρακαλώ, και αργά. Και τώρα ξεκινάμε τη συζήτηση με τον κύριο Σόλτς. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά, κύριε Σόλτς. Mr. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω δύο λόγια σήμερα εδώ και αναφερθώ στα όσα μας απασχολούν από κοινό σήμερα. Όλοι γνωρίζουμε πως η κρίση του COVID-19 είναι μια πρωτόγνωρη πρόκληση και οι οικονομικές αλλά και οι κοινωνικές επιπτώσεις της θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε έναν κατακαιρματισμό. Και αυτό το γνωρίζουμε και από σημαντικά προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν ε, είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε επιλέξει μια διαφορετική άγουσα σε αυτή την κρίση. Η Ευρώπη λοιπόν ανταποκρίθηκε σε μια τέτοια ιστορική ε, πρόκληση με ε, τα κατάλληλα μέτρα και πραγματικά προέβη σε μια αλληλέγγυα πράξη η οποία μας βοηθάει στο σύνολο της Ευρώπης αλλά και αυξάνει το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίω. Οπότε σας ευχαριστώ ε, σας ως Ευρωβουλευτές που μου δίνετε, μου δίνετε δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση και αναφερθώ ε, στη συνεργασία μας ακριβώς και στο τι κάνουμε από κοινού. Η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη είναι σοβαρή και γι' αυτό είναι ε, σημαντικό σε αυτό το δεύτερο έμεση του 2020 να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να ανακάμψουμε λίγο από αυτήν την σημαντική οικονομική ύφεση. Οι τελευταίοι δείκτες μας ε, μας δείχνουν ότι υπάρχει ελπίδα για μια ανάκαμψη σε μια σειρά από κράτη-μέλη και για το σύνολο της Ευρώπης το βλέπουμε, αλλά οι εξελίξεις αυτές παραμένουν αβέβαιε και δεν μπορούμε ε, σε καμία περίπτωση να πούμε ότι έχουμε πραγματικά ξεπεράσει οριστικά την κρίση. Και βέβαια ο αριθμο των κρουσμάτων παραμένει μια σε πρόκληση και θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Και θα συνεχίσουμε βέβαια να αναπτύσσουμε θεραπείες ε, και εμβόλια. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να επιστρέψουμε ε, στο μέλλον, στην, στο, στην κατάσταση στην οποία βρισκόμασταν πριν από την κρίση. Μια κρίση η οποία βέβαια έχει κοστίσει ακόμα και τη ζωή σε κάποιου συνανθρώπου μα. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα. Το σύνθημα τη Γερμανική Προεδρία του ε, Συμβουλίου είναι μαζί για την ανάκαμψη τη Ευρώπη. Γιατί πραγματικά θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε η Ευρώπη να αντιδράσει και να εξέλθει από την κρίση του COVID-19 ισχυρότερη και δικαιότερη αλλά και πιο βιώσιμη. Εδώ λοιπόν έχουμε νομοθετικές διαδικασίες οι οποίες ε, τρέχουν ειδικότερα σε ό,τι αφορά ε, την, ε, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Next Generation EU προκειμένου ο στόχο μα είναι να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη αυτού του έτου και να ξεκινήσει η εκλογή των κοντιλίων από τον Ιανουάριο του 2021. Θα πρέπει βέβαια για αυτόν τον λόγο να εγκριθούν και σχετικέ νομοθετικέ πράξει. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την απόφαση των ιδίων πόρων αλλά και τι εθνικέ διαδικασίε κύρωση. Ε, το πακέτο λοιπόν ανάκαμψη μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανθεκτικότητα και στην ανταγωνιστικότητα των εθνικών μα οικονομιών και επίση είναι στρέφεται προς το μέλλον γιατί μπορεί να υποστηρίξει και την, τον ψηφιακό αλλά και τον οικολογικό μετασχηματισμό. Και γι' αυτό βέβαια ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο έτσι ώστε να ε, λάβουμε βράχη πρόθεσμα μέτρα μέσω μεταρρυθμίσεων και μέσω επενδύσεων αλλά και μέσω πρόθεσμα να μπορέσουμε να προωθήσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, με το ε, πακέτο ανάκαμψης ε, θέλουμε και επιτυχάνουμε ήδη ένα νέο επίπεδο κοινή δημοσιονομική πολιτική, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία έτσι ώστε να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο την ολοκλήρωση αυτή τη δημοσιονομική πολιτική. Τώρα, τα απαραίτητα κονδύλια ω Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα αντλήσουμε από, κοινού στις, από τι αγορέ και βέβαια θα τα εξοφλήσουμε από κοινού. Και γι' αυτό θα, ήδη θα πρέπει από τώρα να αρχίσουμε να σκεφόμαστε πώ μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα τα κοινά μας έσοδα και εδώ αναφέρουμε ιδιαίτερα στους ε, ίδιους ε, πόρους, για παράδειγμα το πώς ε, μπορούμε να έχουμε καλύτερη διαχείριση για παράδειγμα και των εσόδων από το σύστημα εμπορίας εκπομπών και την διεύρυνσή του και στις, στην αεροπορία και στην αυτιλία, αλλά και με το μηχανισμό συνορική προσαρμογή άνθρακα, το ε, border ε, mechanism, αλλά και το πώ, για παράδειγμα, μπορούμε να ε, θεσπίσουμε και αυτόν τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και να τον συμπεριλάβουμε σε αυτού του πόρους. Ε, βέβαια, ακριβώς όλα αυτά τα ζητήματα ε, δημιουργούν και την κατάλληλη ανάγκη για περαιτέρω συζήτηση όπως θα πρέπει να γίνει και στο Συμβούλιο. Πάντως η κρίση και ε, το πώς αντιδράσαμε σε αυτή ε, καθιστούν ένα γεγονό σαφέ ότι χρειαζόμαστε ένα κοινωνικό σύνολο το οποίο θα πρέπει να έχει το κατάλληλο εξοπλισμό, τα κατάλληλα μέσα στη διάθεσή του και να λαμβάνει και δράση. Και γι' αυτό σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να συμμετάσχουν με δίκαιο τρόπο στα φορολογικά έσοδα. Έσοδα, έσοδα τα οποία θα μα επιτρέψουν βέβαια να υποστηρίζουμε και να προστατεύουμε τις επιχειρήσει μας και τους πολίτες μας. Και το, ε, πόσο σημαντικό είναι αυτό μας το καταδεικνύει και η ψηφιοποίηση η οποία βέβαια ε, δημιουργεί ε, και μεγάλες αλλαγές σε ό,τι αφορά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και την δομή τους. Και υπάρχουν λοιπόν για παράδειγμα πολλά παραδείγματα τέτοιου είδους επιχειρήσεων οι οποίες είναι πολύ επιτυχημένες αλλά οι οποίες ε, συμβάλλουν ελάχιστα ακριβώ στα φορολογικά έσοδα. Και για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση μπορούμε να έχουμε μια συντονισμένη δράση εδώ και επιχαίρω το γεγονό ότι ε, και στον ΩΣΑ γίνεται μια ε, ε, πολύ καλή δουλειά προκειμένου ακριβώ να συντονίσουμε ε, διεθνώς ε, την φορολόγηση αυτών των ε, online πλατφορμών και προκειμένου να έχουμε μια αποτελεσματική φορολόγηση επιχειρήσεων. Πρόκειται λοιπόν για προσπάθειες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και τις οποίες λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Εδώ το ζητούμενο είναι μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική για μια δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση και εδώ έχουν υποβληθεί μια σειρά από προτάσεις και θα υποβληθούν και περαιτέρω προτάσεις. Εδώ για παράδειγμα αναφέρομαι στο ζήτημα της ενοποιημένης ε, φορολογικής βάσης επιχειρήσεων και τις σχετικέ προτάσεις ε, της Επιτροπής, αλλά και προτάσεις από ορισμένα κράτη-μέλη όπως για παράδειγμα η Γαλλία και η Γερμανία. Από εκεί και μετά θέλουμε να ενισχύσουμε περισσότερο την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μα εδώ. Δύο σημαντικά ζητήματα εδώ είναι καταρχήν η ε, Τραπεζική Ένωση και από και η ε, Ένωση των Κεφαλαίων Αγορών. Ε, πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε αυτέ τι ενώσει έτσι ώστε να έχουμε και μια, μια σημαντική πρόοδο για την οικονομία μας. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις εθνικές οικονομίες των κρατών Και στο πλαίσιο της δικής μας προεδρίας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε και αυτή την πτυχή. Θα πρέπει δηλαδή να γίνουν και σχετικέ συζητήσει, για παράδειγμα μεταξύ άλλων και για την οριστικοποίηση τη συμφωνία Βασιλεία 3 με βάση τη σχετική πρόταση τη επιτροπή. Σημαντική, σημαντικός είναι και ο ε, ψηφιακός μεταχειρισματισμός για μας στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ε, δηλαδή είναι ένα ζήτημα ε, στο οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα τεχνικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε να προστατεύσουμε την σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των αγορών μας, αλλά προστατεύοντας ταυτόχρονα και τα συμφέροντα των πολιτών μας. Εδώ αναφέρομαι ιδιότερα σε κάποια κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και πιο συγκεκριμένα ε, το ζήτημα των stable coins. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν εδώ πολύ επικριτικές απόψεις και υπάρχουν και πολύ σημαντικές Αποφάσει που ήδη διατυπώνονται από την πλευρά όλων των εμπλεκόμενων φορέων εδώ στην ε, Ευρώπη και νομίζω πως είναι σωστό αυτό γιατί θα πρέπει να κάνουμε ε, ό,τι μπορούμε και προκειμένου να μην αναλάβουν κάποιοι ιδιωτικοί φορεί στο μέλλον ε, αρμοδιότητε οι οποίε ε, μέχρι τώρα ασκούνται από δημόσιου φορεί. Επίση, θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε περιττέρω πρόοδο σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο. Χρειαζόμαστε λοιπόν εδώ μια αποτελεσματική εποπτική δομή σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ε, προστατεύσουμε την ακαιρεότητα των κεφαλαίων αγορών. Και εδώ θα υπάρξουν, θέλουμε να υπάρξουν και συμπεράσματα του Συμβουλίου σε συνέχεια των σχετικών προτάσεων τη Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα, και εδώ μπορεί να συμβάλλει ο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ε, θέλουμε δηλαδή να προωθήσουμε τι σχετικέ προσπάθειε που γίνονται. Έχουμε ήδη συμφωνήσει επί μια ταξονομίας σε ό,τι αφορά ακριβώς τον βιώσιμο χρηματοπιστωτικό τομέα και μέσα στον επόμενο ε, μήνα θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας σε ό,τι αφορά τη διατύπωση συγκεκριμένων κριτηρίων screening ε, και για τον καθορισμό των του ποιε είναι εκείνε τι δραστηριότητε που μπορούν να γίνουν αντιληπτέ ω βιώσιμε. Και από εκεί και μετά, βέβαια, θέλουμε να υποστηρίξουμε και τη δημοσίευση τη ανανεωμένη στρατηγική για, για την βιώσιμο χρηματοπιστωτικό τομέα. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε πολλά ακόμα, αλλά θα περιοριστώ σε αυτά και αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα κάνουμε. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σόλτς, περνάμε στη συζήτηση να υπενθυμίσω σε όλα τα μέλη ότι έχουμε δύο λεπτά για τις ερωτήσεις και τρεις, τρία για τις απαντήσεις. Και ξεκινάμε με τον κύριο Μάρκος Φέρμπερ από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίαση. Χαιρόμαστε φυσικά ως ΕΛΚΑ που θα έχουμε μια στενή συνεργασία μαζί σας και με το Ίδρυμα Ρόμπερτ Κοχ, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να συναντιόμαστε κιόλα. Έχω δύο θέματα. Πρώτον, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αναφέρατε, είναι μια προτεραιότητα η χρηματοδότηση της καταπολέμησης του ξεπλήματος μαύρου χρήματος και της τρομοκρατίας. Με, την, ε, ε, με τον γερμανικό ΣΔΟΕ ε, έχουμε την εμπειρία ότι δεν είναι οργανωμένη το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. και υπήρξαν ε, κάποιες υποψίες μάλιστα ε, για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τιμωρήθηκαν και γι' αυτό. Πώς βλέπετε να οργανώνεται στο μέλλον η, καταπολέμηση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Επίσης ε, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή χρεώνεται. Η καγκελέρος είπε ότι γίνεται για μια φορά με συγκεκριμένο σκοπό. και είπε και δημοσίες ότι πρόκειται για μια χρηματοδότηση που αποτελεί πραγματική πρόοδο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε που, σε τι έγκυται αυτή η πρόοδος. Δεν θέλουμε να γίνουμε μια ένωση χρέους. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, πρώτον για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Ε, τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει πολύ η Γερμανία με διαφορές διαδικασίες ε, και έχουν υπάρξει και πολλές αποφάσεις που υποστηρίζουν ώστε η Financial Intelligence Unit που έχει αλλάξει ελάχιστους υπαλλήλου, έχει δραστηριοποιηθεί πολύ σε συνεργασία με την αστυνομία και έχουν ε, ε, συμβάλει πολύ μαζί με τις τελωνικές αρχές που έχουν πολλές επιπλέον δυνατότητες. Έχουμε τεράστια αύξηση προσωπικού και φυσικά η βάση είναι ότι ε, υπάρχει και αντίστοιχη επιτυχία. Υπάρχει εξοπλισμός τεχνικός και τεχνολογικός που βασίζεται και στο γεγονός ε, ότι έχουμε στοχευμένες ε, ε, δράσεις βάσει πληροφοριών που λαμβάνουμε μέσω τεχνικών διαδικασιών και αναλύσεων και άλλων μέτρων. Η τεχνολογική ικανότητα δεν υπάρχει μόνο στα χέρια ορισμένων μόνο που πραγματοποιούν ξέπνομα μαύρου χρήματο ή παρανομή οικονομία, αλλά και σε άλλους που ασχολούνται με τεχνική νοημοσύνη και χρησιμοποιούν και άλλα μέσα ούτω ώστε έτσι να μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν ληφθεί υπόψη. Επιπλέον υπάρχει ευρεία νομοθέτηση. Υπάρχουν περισσότερες αρμοδιότητες δράσης. Κατά την απόψη μου δεν έχει κλείσει, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ακόμα. Σημαίνει και την πρόσβαση ορισμένων αρχών στα ίδια δεδομένων. Ε, ένα θέμα που επίσης ε, οδηγεί σε συζητήσεις είναι αναγκαίο να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατότητες ε, σε όσους εργάζονται στον τομέα. Είμαι πεπισμένος ότι δεδομένη της παγκόσμιας προσπάθειας θα καταφέρουμε και στην Ευρώπη να συνεργαστούμε καλά και αν γίνουν σωστές ε, ε, προτάσεις για τις εποπτικές αρχές στην Ευρώπη θα μπορέσουμε να βρεθούμε σε θέση ώστε να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο καταπολέμησης της νομοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όσον αφορά το ερώτημα του πώς μπορούμε να ανακάμψουμε στην Ευρώπη θα εξαρθεί από διάφορες αποφάσεις που θα ληφθούν φέτος, τις οποίες εγώ υποστηρίζω. Πρώτον, οι δέσμε μέτρων που παρουσίασαν οι Υπουργοί Οικονομικών από την αρχή της κρίσης σχεδόν 540 εκατομμυρίων ε, ευρώ με τις επιστώσεις ε, για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη Κάτι που ορισμένε χώρε λόγω τη δική μου ε, τραπεζική δομή μπορούσαν να το κάνουν, αλλά άλλε όχι. Γι' αυτό είναι σημαντικό και εδώ να δημιουργήσουμε ε, ένα level playing field, ίσες συνθήκες ε, για όλους στην Ευρώπη. Αυτό ισχύει και για το πρόγραμμα SUR που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χρήματα για τη μερική ανεργία, ώστε να, να επιχειρήσει στην Ευρώπη και τα επιπλέον, επιπλέον πιστώσει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Η δεύτερη απόφαση είναι τα μέτρα που έχουν να κάνουν με το recovery program, με το πρόγραμμα ανάκαμψης που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί με τους υπόλοιπους και εγώ έχω επιμείνει πολύ ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση και ζήτησα να προχωρήσουμε προς το αποτέλεσμα το οποίο ε, φτάσαμε να υπάρχουν ε, πιστώσεις δάνεια ούτως ώστε να υποστηριχθεί η δραστηριότητα των ε, κρατών ε, σε θέματα όσον αφορά την κρίση του κορώνα. Μιλάμε για ε, άμεση βοήθεια αλλά και έμεσα μέσω των προπολογισμών των κρατών. Έχει να κάνει πάντα με την ανάκαμψη. Η διαδικασία λοιπόν έχει θεσπιστεί όπως έπρεπε. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη πρόοδος και είμαι ειδικότερα της άποψης ότι αυτά τα κονδύλια τώρα πρέπει να πάνε εκεί που βρίσκεται η κρίση. Τώρα που λαμβάνει η χώρα η κρίση και όχι αργότερα, γιατί είναι πραγματικά μια πολιτική αντιμετώπιση τη κρίση. Είναι σαφέ ότι όποιο παίρνει ε, δάνεια πρέπει να τα ε, εξοφλήσει, να τα επαναπληρώσει. Αυτό προβλέπεται. Ήδη βρισκόμαστε τώρα στην αρχή του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και αυτό θα ξεκινήσει τώρα. Και ε, το ερώτημα είναι από πού. Και η σαφή απάντηση είναι ότι ε, μια τέτοια αντιμετώπιση κρίσης ε, με τη λήψη ε, δανείων έχει μια ιδιαίτερη διαδικασία μέσω των ιδίων πόρων θα πρέπει να καλυφθούν αυτά. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πτυχές, υπάρχει μια διαβούλευση και θεωρώ ότι είναι μια καλή διαδικασία που θα βοηθήσει την Ευρώπη να ενισχυθεί. Ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Χωνος Φερνάντες σοσιαλδημοκράτες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ Σόλτς, που είσαστε εδώ. Σίγουρα θα συνεργαστούμε τους επόμενους μήνες πολύ καλά και για φακέλους που δεν έχουν καν ανοίξει ακόμα. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, τον Ιούλιο που μας πέρασε καλωσορίσαμε την συμφωνία του Συμβουλίου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όμως υπήρχε και το θέμα της ανάκαμψης. Και εκεί οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι αποφάσεις που εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για το περιθώριο ελιγμών που υπάρχει προκειμένου να διαπραγματευτεί το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο για το χρηματοδοτικό αυτό μέσο. Ξέρετε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για αυτό το εργαλείο βρίσκεται στα χέρια του Συμβουλίου. Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια διαφορετική άποψη και θέλουμε να καταλήξουμε πριν από τα τέλη της χρονιάς. Γι' αυτό λοιπόν ρωτάω, πώς θα διαχειριστείτε την κατάσταση εσείς και αν θα μπορέσετε να πείσετε τους συναδέρφους σας στο Συμβούλιο να αλλάξουν στάση. Δεύτερον, όσον αφορά για το μέσο στήριξη τη φερεγγιότητα. Όπω γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να διαγράψει αυτή την πρωτοβουλία. Εμεί όμω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δουλεύουμε πάνω σε αυτή την πρόταση και δεν ξέρω αν βλέπετε κάποια δυνατότητα να διατηρηθεί αυτή η πρόταση ζωντανή. Γιατί τελικά είναι μια από τι πιο σημαντικέ πρωτοβουλίε προκειμένου να διατηρηθεί μια ισότιμη σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων απέναντι στην πανδημία. Ευχαριστώ. Please Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά καταρχήν το ζήτημα που θέσατε, σε ό,τι αφορά το σε δημοσιομερικό πλαίσιο αλλά και το μηχανισμό ε, ανάκαμψη και ανθεκτικότητας, ε, δηλαδή όλα όσα έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο του πακέτου Next Generation EU, να πω ότι ναι, προφανώς όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν και γνωρίζετε πως έχουν γίνει εδώ πολλές προσεκτικές διαπραγματεύσεις, ε, ε, πολλά διαφορετικά συμφέροντα υπήρξαν εδώ που έπρεπε να συντονιστούν μεταξύ τους. Υπάρχει βέβαια και αυτή η αλεξάρτηση μεταξύ πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και Next Generation EU, οπότε ακριβώς επειδή δεν μπορεί να διαχωριστεί κανένα από αυτά τα στοιχεία, από τα υπόλοιπα, δεν θα πρέπει και να το ξεχνούμε αυτό όταν τα συζητάμε ήταν πολύ δύσκολο και πολύ περίπλοκο να φτάσουμε σε μια συμφωνία ως προς το πώς ακριβώς τα επιμέρους προγράμματα θα πρέπει να προωθηθούν και προφανώς όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτές τις διαπραγματεύσεις συνεχίζουν να υπερασπίζονται τα δικά τους συμφέροντα, τη δική τους θέση. Και βέβαια θα χρειαστούμε κάποιο ακόμα χρόνο για να καταλήξουμε εδώ οριστικά, αλλά ε, σε κάθε περίπτωση νομίζω πως ο στόχος ε, όλων είναι να φτάσουμε έως τα τέλη του χρόνου σε οριστική συμφωνία έτσι ώστε από τις αρχές του επόμενου χρόνου να αρχίσει η εκταμείευση των σχετικών κονδυλίων. Γιατί πρόκειται για κονδύλια τα οποία χρειάζονται πολλά κράτη-μέλη και νομίζω πως ε, θα αποτελούσε και ένα πολύ θετικό μήνυμα για την παγκόσμια οικονομία, το να είναι δηλαδή έτοιμη αυτή η συμφωνία μέχρι τα τέλη του χρόνου. Σε ό,τι αφορά τώρα το ε, δεύτερο ε, ερώτημα που θέσατε, ε, δεν το κατάλαβα καλά από τη διερμηνία. Ίσως θα μπορούσατε να μου το θέσετε στα αγγλικά ε, για να είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα τι με ρωτήσατε. Maybe, Jonas, you can repeat the question. Μπορείς να επαναλάβεις την ερώτηση, Γιώνας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι ίδιες ήτανε. Το πρώτο ήταν όσον αφορά την ανάκαψη και την ανθεκτικότητα, ότι το Κοινοβούλιο έχει μια διαφορετική θέση και θα πρέπει να διαπραγματευτούμε. Και η δεύτερη ερώτηση είχε να κάνει με τον μηχανισμό στήριξης φερεγγιότητας. Ja, Danke für die, das Solvency Support Instrument, das war ja die Frage. Ναι, αυτό είναι το ερώτημα που δεν είχα καταλάβει το Solvency Support Instrument, νομίζω πως αποτελεί ναι τμήμα του συνολικού πακέτου και νομίζω πως μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω με βάση το, το βασικό σκελετό του, όπως ε, αν θέλετε αυτό εγγραφήθηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Οπότε αν με ρωτάτε κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει ναι να συνεχίσει η, η δουλειά που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, ναι θεωρώ πως θα πρέπει να συνεχίσει. Chair, do you wish to proceed? Πρόεδρε, θέλετε να συνεχίσετε. Hello? Please go ahead, Chair. Παρακαλώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, είχα αποσυνδεθεί για λίγο. Ζητώ συγγνώμη. Δίνω τώρα το λόγο στον Λουίς Γκαρικάν από το Ρινιού. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι ο συντονιστής του Renew Europe, ε, κύριε Σόλτς, και θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τις προσπάθειες που έχετε κάνει εσείς, κύριο και ο κύριος Βαϊτσάκερ, για να μπορέσετε να φτιάξετε ένα πρόγραμμα ανάκαμψη ε, φιλόδοξο που μα βοηθά να βγούμε δυνατότερα από την κρίση. Υπήρξε μεγάλη επιτυχία μαζί με την καγκελάριο φυσικά. Έχω δύο ερωτήσει. Πρώτον, για το χρονοδιάγραμμα των ιδίων πόρων. Είπατε ότι συμφωνείτε ότι χρειάζονται ήδη οι πόροι, αλλά το Κοινοβούλιο αυτό ανησυχεί για τη δέσμευση του Συμβουλίου στον αφορά του ίδιου πόρου. Η γλώσσα που συμφωνήσατε δεν δείχνει ισχυρή δέσμευση. Σερνόμαστε ουσιαστικά χωρί να καταλήγουμε σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Ο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών έχει αντίσταση. Δεν αναφέρεται την CCTV σε γλώσσα έτσι του Συμβουλίου. Εσείς λέτε δεν σε αρέσει το ETS ως ιδιοσπόρος, ενώ είναι ένα από αυτά που εμείς στο New Europe θεωρούμε τα πιο λογικά. Πόσο ε, αξιόπιστο είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα αυτό για τους ίδιους πόρους και πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί. Θέλω να ακούσω επίσης ε, το, είναι άποψη για το μέλλον των δημοσιονομικών κανόνων ε, τη Ένωση Θέλουμε όλη η οικονομική σταθερότητα και εσεί, αλλά το θέμα είναι ότι οι κανόνε αναβάλλονται και θα είναι δύσκολο να ξαναπάμε στου ίδιου παλιού κανόνε του Μάστρεχτ. σαφώ το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη, ε, με εστίαση σε κάποιε ζημίε και σε κάποια ελλείμματα είναι κακό οδηγό για μια μελλοντική πολιτική συμφωνία με τη σύσταση ε, το να μεταρρυθμιστεί το Σύμφωνο Σταθερότητα Ανάπτυξη και ποιε είναι οι απόψει για το πώ θα πρέπει να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ. Όσον αφορά τους ίδιους πόρους, είναι κεντρικό κομμάτι των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Είμαι αισιόδοξο ότι θα υλοποιηθούν για να διευκρινίσω λίγο για αυτή τη συγκεκριμένη κρίση. Για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσαμε ειδικότερα για το ε, τα 2021, 2022 και 2023 ε, να κινητοποιήσουμε περαιτέρω κονδύλια ούτως ώστε να σταθεροποιηθούν οι οικονομίες των κρατών μελών και να μεριμνήσουμε ώστε κοινού να έχουμε ανάκαμψη. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ καλό. Ειδικότερα που έχουμε τώρα να λάβουμε και αποφάσεις στο, την οικολογική ε, μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν θα παραμείνουν έτσι αυτά τα χρέη, πρέπει να εξοφληθούν. Οπότε ορίστηκαν κριτήρια για αυτό το σκοπό. Γι' αυτό συνδέεται με αυτά ε, η απόφαση για τους ίδιους πόρους. Ε, αλλιώς θα μέναμε χωρίς λύση. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι αισιόδοξο ε, ω πολίτη Ευρώπη για τι μεταρρυθμίσει, ε, υπόσχομαι ότι στο τέλο ε, θα έχουμε μια δράση πολύ ισχυρή, μια νομική πράξη που θα είναι ισχυρή και θα μα βοηθήσει να φέρουμε αποτέλεσμα. Τώρα, αν κάνει τι προσπάθειε και θελήσει να το υποστηρίξει το Κοινοβούλιο, του χρόνου και του παραχρόνου θα βοηθήσουμε την κατάσταση και δεν θα χρειάζεται να λαμβάνουμε νέες αποφάσεις κάθε χρόνο. Τα ζητήματα της ETS, ε για παράδειγμα και η επέκτασή τους στις θαλάσσιες και στις ε, ε, ενέργειε μεταφορές είναι ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί και δεν, υπάρχουν, δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένο καθεστώ από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό είναι πολύ πιθανό να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση όταν θα έχουμε τι τεχνικέ λεπτομέρειε και δεν υπάρχουν αλλακτικοί τρόποι που να μας δίνουν παρόμοια αποτελέσματα. Όσον αφορά το ζήτημα του φόρου για το πλαστικό, δεν φόρος είναι ένα τέλος ε, από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών βάσει στατιστικών στοιχείων για το μη χρησιμοποιημένο πλαστικό. Για πλαστικό δηλαδή που δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Οπότε είναι εύκολος ο φόρος να οριστεί. Τώρα για το ερώτημα της ψηφιακή φορολογία και της φορολογία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Έχω ήδη πει ότι είναι άλλου είδου συζητήσει. Πιστεύω ότι για τη ψηφιακή φορολόγηση θα βρούμε σύντομα και πρέπει να βρούμε μια λύση. Πολλές χώρες ε, της Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποφασίσει να εισάγουν τέτοια φορολόγηση, αλλά ε, ε, απειλούνται με σοβαρέ αντιδράσει αν το κάνουν αυτό Οπότε θα πρέπει ως λύση να έχουμε μια γενική παγκόσμια ε, συμφωνία που θα δούμε αυτό το φθινόπωρο. έστω να υπάρξει ένα blueprint για αυτό το θέμα. Είναι θέμα που αφορά τον ΩΣΑ ε, και εμάς. Όσον αφορά τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είμαι πεπισμένο ότι έχει λόγο ύπαρξη. Οι χώρε που υπάρχει τέτοιο φορό ή που έχουν αποφασίσει να εισάγουν τέτοιο φόρο ε, ε, η Γαλλία ας πούμε είδε ότι στο σύστημα που έχει η Γαλλία σχεδόν το 90% των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα μπορούσαν να φορολογούνται με αυτό το γαλλικό σύστημα. Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ίδιο πόρο με θετικά αποτελέσματα και για την ελληνική στην Ευρώπη. Ορισμένες χώρες θα ε, έχουν περισσότερα έσοδα, θα επωφελεί όλους Ε, οι χώρε λοιπόν που δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά για ποιο λόγο πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το φόρο, ε, γιατί θα έχουν χαμηλό εισόδημα, θα το καταλάβουν ε, όταν εστιαστούμε για να εξηγήσουμε το αλληλέγγυα διάσταση. Οπότε θέλουμε να το υπογραμμίσουμε τη σημασία. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κοινοί δημοσιονομικοί κανόνες. Πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε ε, πριν τελειώσει το φετινό έτος ε, να καταλάβουμε ότι είμαστε σε μια δύσκολη ε, κατάσταση και πρέπει να δράσουμε αμέσω. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κούνερ τώρα το λόγο. ID. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, Ευχαριστούμε ε, κύριε Υπουργέ. Αναφερθήκατε ε, στο ε, πακέτο ανάκαμψη ω κάτι πολύ σημαντικό για όλα τα κράτη-μέλη και για τη Γερμανία. Και είπατε ότι είστε βέβαιος ότι η κοινή άνεψη δανείων θα είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Οι ε, γερμανικοί μισθοί βέβαια ε, βρίσκονται λίγο ανώτερα, από, είναι σε πιο υψηλά επίπεδα από τον μέσο όρο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η φορολογική επιβάρυνση αυτών των μισθών είναι υψηλότερη από τις υψηλότερες στον κόσμο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ουσιαστικά έχει διατηρήσει πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια ταυτόχρονα τα ενίκια παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά, τα οποία ε, για παράδειγμα βρίσκονται στο ίμιση των ε, σχετικών ενικίων σε άλλες χώρες όπως η Ιταλία για παράδειγμα, η Ισπανία και άλλες χώρες. Βρίσκονται πολύ χαμηλότερα δηλαδή από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ουσιαστικά λοιπόν η Γερμανία είναι μια χώρα πλούσια με πολλούς φτωχούς ε, πολίτε. Τα περισσότερα λοιπόν από τα κονδύλια για την αντιμετώπιση τη κρίση θα πάνε προ τον νότο τη Ευρώπη ενώ η, ε, η Γερμανία παρότι συμμετέχει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή την χρηματοδοτική υποστήριξη θα λάβει πολύ λίγα από αυτά τα κοντήλια Γιατί λοιπόν θα πρέπει ε, σε βάρος Γερμανών πολιτών οι οποίοι πραγματικά έχουν οικονομικά προβλήματα να επωφεληθούν ε, πλούσιοι πολίτες από χώρες του Νότου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο κύριος Σόλ, σας ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα η δική μου απάντηση μπορεί να είναι σύντομη και περιεκτική σε αυτό που είπατε. Δεν νομίζω πως ε, μπορεί κανείς ε, να παραβλέψει τα όσα προκύπτουν από, ε, από μια εθνική οικονομία. Η Γερμανία πραγματικά είναι, έχει μια ισχυρή οικονομία με ισχυρά έσοδα. Και αυτό ισχύει για τη Γερμανία και για τους πολίτες της. Ό,τι και αν πει κανείς ε, και όποια άλλα στατιστικά και αν χρησιμοποιήσει δεν μπορεί τελικά να, να κλονίσει μια τέτοια αλήθεια όπως είναι το γεγονός ότι δηλαδή η Γερμανία έχει μια ισχυρή οικονομία. Τώρα αν θέλει κανείς να βρει κάποιον αργόριθμο για να ε, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τελικά η Γερμανία από τις φτωχές χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι να πω, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι προσβλητικό και για την νοημοσύνη μας. Νομίζω πως όλοι γνωρίζουν ε, ότι αυτό που μόλις τώρα είπατε δεν ισχύει. Πέραν αυτού, είδαμε ε, ότι η Γερμανία διαθέτει και έναν πολύ ισχυρό δημόσιο τομέα υγείας. Ε, έχει ένα υψηλό αριθμό, για παράδειγμα, νοσοκομειακών κλινών και ακριβώς αυτή η δυνατότητα ε, και αυτό ο ισχυρό δημόσιο τομέα υγεία μα επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε με σχετικά αποτελεσματικό τρόπο την πανδημία και τι οικονομικέ επιπτώσει τη νύχη. Άρα λοιπόν δεν συμφωνώ με την άποψή σα. Κάνετε λάθο. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, Σβέν Κίγκολτ, από τους Πράσινους, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, καλώς όρισατε πρώτα απ' όλα. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπουμε εδώ στην Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Οικονομικών ε, για το ρόλο που έπαιξε υπό τη δική σας ε, καθοδήγηση για το σχέδιο αυτό προϋπολογισμού και τα σχέδια για το Ταμείο Ανάκαμψης. Λύσατε περισσότερα προβλήματα από ότι η πλειοψηφία αυτού του Κοινοβουλίου ε, από την και στο πλαίσιο των ε, προπολογισμού ε, ακόμα συζητούνται αυτά τα θέματα. Πρέπει να το πούμε καθαρά εδώ ταυτόχρονα. Βλέπουμε ότι στην κρίση του κορονοϊού πόσο σημαντική είναι η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλοί στην οικονομία και στην κοινωνία υποφέρουν σοβαρά. Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν κερδίσει κάποιες ψηφιακοί όμιλοι όπως το Amazon σε σχέση με, τους, ε, με τα καταστήματα. Τα τοπικά καταστήματα έχουν ε, επωφεληθεί υπερβολικά από την κρίση και ε, δεν φορολογούνται ακόμα σωστά. Το κοινοβούλιο εδώ προτιμά ε, να υπάρχει σωστή φορολόγηση και των μεγάλων επιχειρήσεων και των ψηφιακών επιχειρήσεων. Γι' αυτό σας ρωτάω. Δύο χρόνια αφού εδώ μιλήσατε, προειδοποιείτε για την φορολογική διαφάνεια, είστε εδώ προσωπικά και είστε υπέρ. Τι θα γίνει με το Συμβούλιο με αυτό το θέμα, ούτως, αφού ε, η Γερμανία δεν συμφώνησε με την τελευταία πρόταση της Φιλανδίας, πότε θα υπάρξει αυτή η φορολογική διαφάνεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πότε η Προεδρία του Συμβουλίου θα οργανώσει μια νέα ψηφοφορία. Και το ίδιο ερώτημα έχω και για τον, για τον ψηφιακό φόρο. Αυτός ο ψηφιακός φόρος ο οποίος καθυστερεί και έχουμε χάσει ήδη 10 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη εξαιτία αυτού, 10 δισεκατομμύρια ευρώ, πότε θα τεθεί στην ημερήσια διάταξη. Αυτό το κοινοβούλιο έχει αποφασίσει θετικά και περιμένουμε το Συμβούλιο των κρατών μελών υπό Γερμανική Προεδρία να λάβει και τη σχετική απόφαση. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Αυτή τη στιγμή σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο στην Ευρώπη με τα δύο μεγάλα καθήκοντα που έχουμε να εφαρμόσουμε ε, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο το πολιτισμο δημοσιονομικό πλαίσιο και το μέλλον της Ευρώπης με το Ταμείο Ανάκαμψης. Όσον αφορά το country by country reporting, ε, πράγματι χρειαζόμαστε μια απόφαση για αυτές τις εκθέσεις αναχώρα. Πριν δύο χρόνια, ξέρω ότι δεν είπα αυτό που συνοψίσατε εσείς εδώ, αλλά έθεσα το ζήτημα του τι είναι υπέρ και τι είναι κατά στη γερμανική κυβέρνηση. Όπως ξέρετε αυτό το ερώτημα δεν έχει βρει σαφή απάντηση. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα ενδεχομένως καλό εργαλείο και τώρα η κατάσταση στην Ευρώπη θα εξαρτηθεί από το κατά θα μπορέσει να συμφωνηθεί. Σε κάθε περίπτωση έχω την εντύπωση ότι η πεποίθηση ότι είναι σημαντικό ε, γίνεται όλο και πιο βέβαιη. Τώρα όσον αφορά τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε μια λύση. Έχω πει ήδη ότι ελπίζω να έχουμε το blueprint ε, το φθινόπωρο φέτο στο πλαίσιο του ΟΣΑ και να μπορέσουμε να οργανώσουμε μια ε, παγκόσμια ε, ύπαρξη αυτού του μέσου. Το συζητάμε εδώ πολύ στην Ευρώπη και αυτό θα επηρεάσει, θα έχει συνέπειε και το σύστημα ε, φορολόγησης επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο, αλλά χρειαζόμαστε παρόλα αυτά μια λύση και θέλω να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά Αυτά τα θέματα που αναφέρατε εσείς ε, συνδέονται και με τα άλλα σημεία που αναφέραμε. Είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Φέτος εγώ θα κάνω προσπάθειες να τα καταφέρουμε και σε αυτόν τον τομέα. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε. Επίνγκ τώρα, ECR. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας ε, σε ό,τι αφορά αυτό το συνολικό πακέτο που έχουμε μέχρι τα τέλη του έτους. Ε, πραγματικά πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε, γιατί υπάρχουν μια σειρά προβλήματα μεταξύ αυτών και η σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα το ζήτημα δηλαδή το κράτος δικαίου και τη σχετική ερωσιμότητας. Από εκεί και μετά η διαδικασία ακύρωσης ε, προφανώς θα πρέπει να τρέξει και σε ό,τι αφορά την ε, απόφαση για του ίδιους πόρου, αλλά εδώ έχουμε 50 διαφορετικά ε, κοινοβούλια που θα πρέπει να ακυρώσουν μια τέτοια συμφωνία. Πώς θα τα καταφέρουμε όλα αυτά. Και από εκεί και μετά ε, να ρωτήσω, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να παρέμβει στις κεφαλαίες προτού ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης από τα επιμέρους κοινοβούλια. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας. Ευχαριστώ, λέω ο Υπουργός, ε, για τα ερωτήματά σας. Θέλω να απαντήσω και στα δύο σκέλη αυτά από κοινό. Γιατί το δεύτερο σκέλος, αν θέλετε, το δεύτερο ερώτημα που θέσατε, υπογραμμίζει το πρώτο. Ναι, είναι σημαντικό να ολοκληρώσουμε ταχαίως και ναι, κατά την άποψή μου θα τα καταφέρουμε ως τα τέλη του έτους. Ναι, Ορισμένε φορέ υπάρχουν προκλήσεις ε, ισχυρές οι οποίες ακριβώς μας ε, επιτρέπουν να επιταχύνουμε διαδικασίες οι οποίες ενδεχομένως για παράδειγμα να χρειαζόντουσαν δύο ή τρία χρόνια για να ολοκληρωθούν. Ε, το ότι είναι δηλαδή σημαντικό αυτό το ζήτημα ακριβώς μας ασκεί περισσότερε πιέσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία στα τέλη του έτου, αντί να επαναπαυθούμε. Σα ευχαριστώ πολύ. τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, με ακούτε, ελπίζω. Δεν ξέρω αν με βλέπετε στην εικόνα. Ευχαριστούμε για την πολύ σημαντική ανταλλαγή απόψεων. Χαίρομαι που βλέπω τόση αισιοδοξία. Υπάρχει και ένα σημαντικό ερώτημα όμως. Ε, για να δούμε τι θέση θα πάρουμε. Η πρόεδρος εδώ είπε για την κρίση του κορονοϊού και πόσο θα αυξηθεί το χρέος εδώ στην Ευρωζώνη. Κατά μέσο όρο, κατά 100% ε, του ΑΕΠ θα αυξηθεί η χρέωση 200% ενδεχομένως η Ελλάδα, 160% η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ιταλία κάτω από το 20%. Η Γερμανία παίζει έναν άλλο ρόλο φυσικά εδώ, πιο κοντά στα κριτήρια του Μάστριχτ φυσικά όσον αφορά το χρέος. Έχει σκεφτεί η Γερμανία ποιε θα είναι οι συνέπειε και για την ίδια ε, για την αντιμετώπιση τη κρίση του κορονοϊού, ποια συγκεκριμένε μεταρρυθμίσει βλέπετε στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, ως γερμανική κυβέρνηση, γιατί φυσικά όταν μιλάμε για τέτοια ποσοστά ε, τα κριτήρια δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα και η Γερμανία ε, έχει μπει σε άλλη οδό ούτως ή άλλως. Και η δεύτερη ερώτηση, επειδή ήθελα πιο συγκεκριμένε πληροφορίε από εσά όσον αφορά το ψηφιακό φόρο και το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ενώ εμεί Μιλάμε για ίδιους πόρους που θέλουμε να δημιουργήσουμε εμείς. Ε, φτιάχνουμε μια κοινή ευρωπαϊκή φορολογική ε, πολιτική που δεν υπάρχει όμως μέχρι στιγμής. Θα βασιστεί λοιπόν σε τι. Ε, ξέρουμε ότι αν δεν υπάρχουν σταθερά θεμέλια τότε οι συμμετοχές των κρατών μελών θα πληρωθούν μέσω του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Το είπατε κι εσείς ε, ότι είναι σημαντική αυτή η διπόρη. Πόσο συγκεκριμένα λοιπόν θεωρείτε ότι μπορούν να υλοποιηθούν αυτοί οι φοροί του ΩΣΑ. Πότε ακριβώς θα υπάρχει, πιστεύετε, ένας ευρωπαϊκός φορολογικός ε, ε, ψηφιακός φόρος. Και δεύτερη ερώτηση. Πώς και πότε θεωρείτε ότι θα υπάρξει φόρος των χρηματόπιστων συναλλαγών. Ευχαριστώ. Πρώτον, ε, θα ήθελα να απαντήσω για το κρατικά χρέη. Έτσι όπως το παρουσιάσετε εσείς στο σενάριο, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους εγώ είμαι υπέρ στις συζητήσεις και στην Ευρώπη και στη Γερμανία του να βρούμε μια λύση με ένα κοινό ταμείο ανάκαμψης. και να το περιλαμβάνει αυτό ε, χορηγίες περισσότερο. Τώρα όσον αφορά τα χρέη των όλων χωρών, ε, όπως το είπατε εσείς, το πρώτο πακέτο των 540 δισεκατομμυρίων που ανέφερα και εγώ και οι πολλές πράξεις αλληλεγγύης μας δείχνουν ότι δεν θέλουμε να αντιμετωπίσει δυσκολίες καμία χώρα να χρηματοδοτηθεί τώρα εν μέσω κρίσης και να ε, επομιστεί όλο το χρέος της ε, ε, ανακάμψη αυτό να γίνει μέσω των κεφαλαίων να χρηματοδοτηθεί και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Μας δείχνει ότι στην Ευρώπη μπορούμε με βιώσιμο και αποτελεσματικό και εύπιστο τρόπο να συνεργαστούμε και να σταθούμε ένα στο πλευρό του άλλου. Αλλά αυτά τα grants φυσικά είναι ένα κομμάτι της απάντησης σε αυτό το ερώτημα. Δεν μιλάμε για χρηματοδότηση προπολογισμού, αλλά συγκεκριμένα μεταρρυθμιστικά έργα. Θα βοηθήσουμε και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίε ε, για να βγουν από αυτές. Τελικά το σενάριο ίσως να έχει άλλη μορφή στο τέλος ε, και όχι μόνο την αλληλεγγύη αυτή που εμείς θεωρήσαμε ότι ήταν απαραίτητη για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Τώρα όσον αφορά το ζήτημα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό και στο μέλλον. Ελπίζουμε να έχουμε κάποια σταθερότητα στο μέλλον. Βασικό κριτήριο όχι μόνο για τη γερμανική αλλά και για την ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, το σημαντικότερο είναι να κάνουμε τώρα ό,τι είναι σωστότερο ώστε να έχουμε καλή έκβαση. Είναι σαφές ότι για να τονώσουμε την ανάπτυξη αυτό πρέπει να γίνει με τα μέσα τα οποία έχω προσπαθήσει να περιγράψω. Τώρα όσον αφορά τους διάφορους ιδιούς πόρους, τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας και το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, για την ψηφιακή φορολογία πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει μια παγκόσμια συνεννόηση για το ζήτημα αυτό. Εμείς έχουμε προσπαθήσει πολύ και ελπίζουμε ότι το φθινόπωρο θα καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Τόσο η Γερμανία όσο και εγώ προσωπικά έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα σαν αυτό που λάβαμε τώρα ως πρόταση από του ευρωπαϊκά κρατημέλη ε, είμαστε τη άποψη ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. η ΕΠΑ συμμετέχουν στις ε, συνομιλίες και οι ΕΠΑ γνωρίζουν ότι δεν συμφέρει κανέναν σε εποχές όπου έχουμε αρκετά προβλήματα με την πανδημία, με τα υγειονομικά, ε, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, με την ανασφάλεια της οικονομικής ανάπτυξης, λόγω των διαφόρων εμπορικών πολέμων, επίσης να μην έχουν προσθεθεί και άλλο πρόβλημα. Ε, να υπάρξουν επαρκή έσοδα λοιπόν ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν ε, όλα τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Οπότε ελπίζουμε να καταλήξουμε σε μια συνεννόηση για το φόρεπτο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ήξερα εδώ και καιρό ότι έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε μια σημαντική πρόοδο Ε, φορολογούμε διάφορα πράγματα στην Ευρώπη και όχι τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγές. Ε, και έχουμε τις δύο μεγαλύτερα χρηματιστήρια του Παρισιού και του Λονδίνου και θα μπορούσε εκεί να γίνει φορολόγηση αυτή χωρίς πρόβλημα. Χωρίς να φύγουν αυτά τα χρηματιστήρια από την Ήπειρό μας. Με το νέο σενάριο των ιδίων πόρων που λέμε ότι χρειαζόμαστε για να επαναχρηματοδοτήσουμε το μεγάλο πακέτο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε για αυτού του φόρους. Είμαι πεπισμένο. Αυτό το πρόβλημα το οποίο παρουσιάσατε υπάρχει έτσι όπως το ε, παρουσιάσετε εσείς χωρίς τους ίδιους ή θα ήταν δύσκολο, αλλά το πρόβλημα είναι και κομμάτι της λύσης. Κανείς ε, δεν θα μπορούσε για δικό του συμφέρον να παρεμποδίσει να καταλήξουμε σε μια απόφαση όσον αφορά του ίδιου πόρου. Είναι απαραίτητη μια τέτοια απόφαση για να κάνουμε τα κοινά βήματα που έχουμε αποφασίσει. Οπότε μερικές φορές η πίεση βοηθά κιόλα την κατάσταση. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Η Λίδια Περέιρα τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σόλτς. Το 2020 είναι το έτος της κρίσης της πανδημίας και πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν στην οικονομική ανάκαμψη προκειμένου η ύφεση να γίνει ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε περισσότερο, να έχουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Πρόκειται για μια πρόκληση αλλά και για μια ευκαιρία να βρούμε νέες καινοτόμε λύσεις και να επιταχύνουμε κάποιες αλλαγές που συζητάμε εδώ και καιρό χωρίς όμως να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα. Όσον αφορά τα δημοσιονομικά βήματα, χαίρομαι για την προσπάθεια που κάνει το Συμβούλιο και η Προεδρία. Ε, φαίνεται ότι η ευελιξία αποτελεί τμήμα της ανάκαμψης και της αντοχής και πρέπει να υπάρχει περιθώριο ελιγμών πράγματι τα επόμενα χρόνια. Τώρα η ερώτησή μου θα επικεντρωθεί στο σχέδιο ανάκαμψης έτσι όπως το σχεδίασε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εσείς πώς βλέπετε την ισορροπία ανάμεσα στις επιχορηγήσεις και τα δάνεια μετά την απόφαση του Συμβουλίου που μείωσε κατά πολύ τις επιχορηγήσεις. Η απόφαση πάντως για την έκδοση χρέους αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Και σε αυτό βοηθάει η απόφαση για τους ίδιους πόρους, η οποία είναι βέβαια μια πρόοδος, αλλά είναι κάπως ασαφής, ενώ χρειάζονται συγκεκριμένες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα για τους ίδιους πόρους, συγκεκριμένα ποιοι θα είναι αυτοί. Τώρα σήμερα η Επιτροπή Προπολογισμών ζήτησε ένα πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων. Η ερώτησή μου λοιπόν προς την Γερμανική Προεδρία είναι ποια είναι η θέση της, ποιο είναι το επίπεδο φιλοδοξίας της για να μπορέσουμε να εισάγουμε μια μεταρρύθμιση για τους ίδιους πόρους. Πιστεύετε ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι ένα παράθυρο ευκαιριών και τι βάση βλέπετε εσείς γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. για το ζήτημα των ιδιών πόρων με ρώτησαν ήδη, οπότε θα προσπαθήσω να επαναλάβω αυτά που είπα. Θεωρώ ότι τώρα χρειαζόμαστε μια ποιοτική ε, μεταβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έρθει με, τα, με τους ίδιους πόρους. Έχει ήδη καταγραφεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου με τη συγκεκριμένη πρόταση για το δέσμι μέτρων για την ανάκαμψη. Το πώς ακριβώς θα γίνει η κατανομή περιγράφεται 90 ε, δισεκατομμύρια grants και τα υπόλοιπα πιστώσεις που θα δοθούν στα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική λύση. Και εκεί τίθεται όλο και περισσότερο το ερώτημα το πώς θα τα καταφέρουμε να, να ληφθεί αυτή η απόφαση για τους ίδιους πόρους. Το περιγράψαν ήδη Κάποιοι ε, συνάδελφοι το είπαν ότι αν δεν τα είχαμε θα ήταν δραματικές οι ε, συνέπειες. Ε, ίσως να χρειάζονται αποφάσεις πιο σημαντικές από ποτέ. Ε, ίσως είναι σημαντικότερο κάπου ότι έχουμε αποφασίσει την ανάκαμψη, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα είναι η ώρα να αποφασίσουμε για τους ίδιους πόρους, παρότι έχουμε στραφεί, είχαμε στραφεί, στρέψει την προσοχή μα σε άλλα θέματα. Την επόμενη εβδομάδα που θα συναντηθούν οι Υπουργοί Οικονομικών θα τεθεί αυτό το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη, ούτω ώστε να συζητηθεί το ζήτημα αυτό. Ο στόχο μου είναι να υπάρξει μια γενικότερη συνείδηση ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τι ημερήσιες διατάξει των τελευταίων χρόνων. Χρειάζεται να δοθεί κάποια συγκεκριμένη πίεση. Ε, η Κομισιόν πρέπει να κάνει ε, προτάσεις, δύο προτάσεις ε, το Μάρτιο του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος, ε, η πρώτη και πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να το αποφεύγουμε, πρέπει τώρα να λάβουμε αυτή την απόφαση, να την προετοιμάσουμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που αναφέρονται στη συμπεράσματα του Συμβουλίου ούτως ώστε να αντικατοπτρίστηκε και κάποια ευρωπαϊκή ποιότητα δεν θέλουμε πόρους από όπου και να έρχονται, θέλουμε οι πόροι αυτοί, ε, από αυτούς τους πόρους να καταλαβαίνει κανείς γιατί είναι ευρωπαϊκά έσοδα αυτά. Δηλαδή πώς έχουν να κάνουν όλη την Ευρώπη και τον ευρωπαϊκό χώρο. Θέλουμε να είναι σαφές ε, ε, και να νομιμοποιείται μέσω από αυτούς η πολιτική που διεξάγουμε στην Ευρώπη και έτσι να γίνουν πρόοδοι στο σχετικό τομέα. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο Κίμ Σούστερ τώρα, Σοσιαλδημοκράτες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που είστε στη διάθεσή μας για τη συζήτηση που κάνουμε ε, και Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που κάνατε εσείς προκειμένου να καταλήξει το Συμβούλιο σε μια συμφωνία τον Ιούλιο ε, σε ό,τι αφορά το σχέδιο ανάκαμψης. Ε, παρά βέβαια όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν αρχικά. Νομίζω δηλαδή πως ε, πραγματικά αυτό που είπατε είναι σωστό. Πρόκειται για μια ιστορική επιτυχία και αποτελεί και μια, ένα ακόμα βήμα προς την δημοσιονομική ολοκλήρωση της Ένωσης. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να αναφερθώ λίγο περισσότερο σε δύο ζητήματα. Νομίζω πως ε, η δημοσιονομική ολοκλήρωση ε, δεν έχει να κάνει με το πώς μπορεί κανείς να κινητοποιήσει περισσότερα κονδύλια, αλλά και η περισσότερη οικονομική σταθερότητα σε ό,τι αφορά ε, ίδιους πόρους, αλλά έχει να κάνει και με το πώς μπορεί κανείς να συντονίσει τις δημοσιονομικές και γενικότερα οικονομικές πολιτικές. Νομίζω πως ε, πραγματικά εδώ υπάρχει περαιτέρω ανάγκη μεταρρύθμισης και η οποία ανάγκη υπήρχε ήδη πριν από την ε, ε, κρίση της πανδημίας. Λόγω δηλαδή και των πολιτικών που ασκούνταν από τα κάστοτε κράτη-μέλη ήταν δύσκολο να προωθηθεί κάτι τέτοιο. Υπάρχει όμως τώρα ο, ο αγώνας κατά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και ο ψηφιακός μεταχειρισματισμός, οπότε θα πρέπει ε, τώρα να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες σε επενδυτικό επίπεδο μέσω μιας σταθερής οικονομικής πολιτικής. Ε, οπότε το ερώτημα που ε, τίθεται εδώ είναι πώς θέλετε εσείς στο πλαίσιο της δικής σας προεδρία του Συμβουλίου να κάνετε μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και πώς θέλετε να εξισορροπήσετε τα διαφορετικά συμφέροντα. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω είναι ε, το γεγονό ότι σε ό,τι αφορά το σχέδιο ανάκαμψη, εδώ στα σχετικά προγράμματα οι δυνατότητε συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ περιορισμένες. Συμφωνείτε ότι θα πρέπει οι αρμοδιότητες συναπόφασης ε, του Κοινοβουλίου θα πρέπει εδώ να ενισχυθούν σημαντικά για παράδειγμα μέσω μια διοργανική συμφωνία. Ποια είναι η δική σα άποψη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, λέει ο Υπουργός, για αυτά τα ερωτήματα ε, και για τα επενετικά σας λόγια. Κατά τη δική μου άποψη είναι ξεκάθαρο λόγω ακριβώ τη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, χρειάζεται να υπάρξει καλύτερο συντονισμό των πολιτικών στι οποίε ε, προβαίνουμε και ακριβώ σε αυτό αποσκοπούν και όλοι οι διάλογοι που διοργανώνουμε. Για παράδειγμα, στο ε, πλαίσιο του επόμενου άτυπου ΕΚΟΦΗΝ θα ε, συζητήσουμε ακριβώς ε, την γενικότερη οικονομική κατάσταση όπως ισχύει ε, και τι θα πρέπει να γίνει από εκεί και μετά. Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή όμως πολιτική, τα βασικά ζητήματα είναι εκεί, εκείνα στα οποία αναφέρθηκα ήδη και δεν θέλω να το επαναλάβω. Παρ' όλα αυτά όμως παραμένουν και κάποιες περαιτέρω αρμοδιότητες και ζητήματα τα οποία μπορούν να μας επιτρέψουν περισσότερη ανάπτυξη επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράδειγμα, αυτό το θέμα της προώθησης Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφάλαια Αγορών είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβάλλει ε, μεταξύ πολλών άλλων στην ε, ε, οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη. Αλλά βέβαια εδώ θα πρέπει να γίνουν προσπάθειε και να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία, γιατί βέβαια δεν έχει κανεί το θάρρο να προχωρήσει σε περαιτέρω προσπάθειε όταν βλέπει ότι ε, μία πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά για την οποία υπάρχει συμφωνία εδώ και δύο χρόνια δεν προχωράει. Επίση, σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη ελάχιστη ε, φορολόγηση των επιχειρήσεων, αποτελεί ένα ζήτημα που μα απασχολεί και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκοσμίω είναι ένα ζήτημα που τίθεται. Ε, δεν μπορούμε δηλαδή εδώ να έχουμε συστήματα αρμπιτρά. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη λύση μεταξύ μα. Ευχαριστώ. Thank the... Σας ευχαριστούμε πολύ. Ερόγλου. Ρινιού παρακαλώ. Yeah. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ Σόλτσα, ευχαριστούμε για την παρουσίαση θα θέλαμε να βρεθεί ο σωστός ε, δρόμος όπως λέτε και σας εύχομαι καλή τύχη φέτος να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα ψηφιακό φόρο για τους μεγάλους ομίλους. Ε, παρ' όλα αυτά έχω μια ερώτηση για τον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τον επίσημο πληθωρισμό του μείον 0,1 υπάρχουν άνθρωποι που την τελευταία δεκαετία ε, ε, φοβούνται για τις συντάξεις τους ε, στα σχετικά ταμεία που με, τους αρνητικούς, με τα αρνητικά επιτόκια φοβούνται ότι θα χάσουν την αξία τους και εκεί θα χάσουν οι άνθρωποι που με τη σκληρή τους δουλειά έχουν δημιουργήσει αυτά τα συνταξιοδοτικά ταμεία και ελπίζαν να διατηρηθούν αυτά για τα παιδιά τους. Οπότε τι θα γίνει με το δημόσιο, θα, αν θα προστατεύσει, θέλουμε να δούμε αν θα προστατεύσει αυτά τα μία. Θεωρείτε ότι ο ευρωπαϊκός ε, ε, προϋπολογισμός ε, μπορεί να βοηθήσει κάπως στη συγκράτηση αυτών των επιτοκίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Θεωρώ ότι για να συζητηθεί χρειάζονται ώρες γιατί είναι πολύ επίμαχο ζήτημα σε οικονομικό επίπεδο. Κατά την απόψή μου δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ήδη από τώρα θα μπορούσε να πει κανεί ότι υπάρχει λόγος να ανισχύει κανεί για, τους, ε, ε, για τα χαμηλά επιτόκια, τα αρνητικά επιτόκια. Είναι τόσο πολύ καιρό που τώρα επανέρχονται σιγά σιγά όχι μόνο στη Γερμανία και στην Ευρώπη αλλά παγκοσμίω και η θέση ε, και μας δείχνει η κατάσταση ότι έχουμε ζήσει με αυτό εδώ και πολύ καιρό και χωρίς κάποιο πρόβλημα και ανεξάρτητα από την πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας ε, υπάρχουν αρκετά χρήματα σε προσφορά. Ε, σε, πολλές, ε, σε πολλά μέρη ψάχνουν οι καταθέτες γρήγορους τρόπους ασφαλής όχι μόνο σε επενδύσεις. Έχουμε ένα πολύ μπανάλ πρόβλημα εδώ. Σε μια χώρα όπως τη Γερμανία η οικονομικά αν θέλαμε να χτίσουμε κάποιο αριθμό σπιτιών, αλλά δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτά από την κεφαλαγορά και χρειάζεται να βρούμε τα χρήματα Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ότι η συντάξη αυτά τα χρήματα θα γίνονταν χαμηλότερες. Ε, στην πραγματική οικονομία χρειάζονται έτσι περισσότερες επενδύσεις. Υπάρχουν και άλλα θέματα που παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά η οικονομική αυτή συζήτηση μας δείχνει ότι αυτό που αναφέρεται δεν έχει να κάνει με τη σημερινή κατάσταση και την πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά παγκόσμιες τάσεις και παγκόσμια οικονομία και θεωρώ ότι μέσω της, ε, των επαρκών επενδύσεων αυτό μπορεί να επιληθεί πρόοδος για την Ένωση Κεφαλαγορών και την Τραπεζική Ένωση πιστεύω ότι δεν πρέπει να υποτιμάται. Θα μας βοηθήσει να έχουμε περισσότερο equity και επενδύσεις στην Ευρώπη. Γιατί σε σύγκριση με τη ΣΥΠΑ οι επενδύσεις για μας είναι 80% πιστώσεις και 20% equity. Ενώ στη ΕΠΑ είναι το αντίστροφο. Και αυτό μας δείχνει ότι με μια κεφαλαιογορά που λειτουργεί κεντρική θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε να προχωρήσουν τα πράγματα και με τις αντίστοιχες συνέπειες φυσικά για το επίπεδο των επιτοκίων. Thank you very much. Uh, very interesting debate. We still have some time, so uh, we have a few requests for Catch the Eye. I give the floor for a two-minute uh, question and answer to eh, Fabio Massimo Castaldo. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο Σόλτ ε, ε, για αυτή την παρουσίαση και για τις προσπάθειες συμβασμού τους τελευταίους μήνες. Θέλω να επιστρέψω σε ένα επιχείρημα που ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι. Θέλω να επενθυμίσω ότι τον Ιούλιο σχεδόν 70 ευρωβουλευτές και μέλη του δικού σας ε, κόμματος των σοσιαλιστών απέθυναν έκκληση ε, προς υποστήριξη του να συμπεριληφθούν στους νέους ιδίους πόρους ο φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Και με ενίσχυση μάλιστα του συντελεστή που συζητείται αυτή τη στιγμή. Και σαφώ, ε, σύμφωνα με αυτά που λέτε, και εσεί συμφωνείτε ότι ο χρηματοπιστωτικό τομέα θα πρέπει να συμβάλλει ε, στο μέγιστο βαθμό ε, δεδομένων των σημερινών συνθήκων. Αλλά το ποσοστό που προκύπτει και βάσει τη γαλλογερμανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικά πολλέ εξαιρέσει. Θα έμεναν έξω και για μένα αυτό είναι πρόβλημα, απαράδεκτο, από τη φορολογική βάση οι συναλλαγέ παραγόγων. Δεδομένου αυτού λοιπόν μειώνονται σαφώς τα φορολογικά έσοδα και δίνεται κίνητρο για την κερδοσκοπία και για επενδύσεις ε, μακροχρόνιες. Ήθελα να μου πείτε εσείς ε, ως ε, εκπρόσωπος γερμανικής κυβέρνησης θα ήθελα να γίνετε λίγο πιο φιλοδοξία. Από το 2012 το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία είναι υπέρ ενός φόρου για όλες τις αγορές, όλους τους φορείς και, όλα τα, και όλους τους τίτλους λόγω της ανάγκης να δημιουργηθούν ήδη οι πόροι για να εγγυηθεί ε, με κάποιο τρόπο η τεράστια προσπάθεια που κάνουμε με το Next Generation EU. Συμφωνείτε μαζί μου ότι το σημερινό μοντέλο λοιπόν που έχουμε υποδιαπραγμάτευση δεν είναι ικανοποιητικό και ότι συνεπώς λόγω της μεγάλης ε, κρίσης υγειονομικής, κοινωνικής και οικονομικής θα χρειαστεί να αυξήσουμε τις φιλοδοξίες μας και να είμαστε πιο φιλοδοξοί και από το μοντέλο που υπάρχει στη γαλλογερμανική πρόταση. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να μπορέσουμε να υπολογίζουμε στη δέσμευσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και τα καλά σας λόγια. Δύο παρατηρήσεις για το ερώτημα αυτό. Πρέπει να πετύχουμε κάτι. Δεν έχει νόημα να αποφεύγουμε ε, πρόοδους διότι δεν φαίνονται πολύ ωραίοι. Πρέπει να καταφέρει κανεί να επιτύχει ό,τι μπορεί να επιτύχει. Και η πραγματικότητα με την οποία έχουμε να κάνουμε είναι ότι οι περισσότερες χώρες ε, ε, που έχουν τέτοια φορολόγηση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, το κάνουν βάσει του γαλλική πρότασης. Οπότε το θέμα είναι τι ακριβώς θα επιτύχουμε. Εγώ θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς το Κοινοβούλιο να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να πιέσει λίγο παραπάνω. Μέχρι στιγμή η συζήτηση για την φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ευρώπη οδήγησε σε ορισμένες ε, χώρες ε, στο αποτέλεσμα ότι γίνεται, ε, στο ότι... Αλλά μα δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες είναι δυνατόν αλλά τα έσοδα λόγω του μεγέθους της ε, κεφαλαγοράς είναι πολύ χαμηλά. Και εκεί τίθεται το ερώτημα του έχει οικονομικό νόημα για όλα τα κράτη-μέλη να κάνουν μια τέτοια μεταρρύθμιση. Και βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς τώρα συζητάμε για το ζήτημα της χρηματοδότησης, της ε, ευρωπαϊκής ανάκαμψης και το ζήτημα του πώ θα παρεμποδίσουμε να επιβαρύνουμε περισσότερο το πολιτιστικο δημοσιονομικό πλαίσιο και η απάντηση είναι ότι μια από τις πολλές δυνατότητες που έχουμε είναι σαφώς ότι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. πολλές χώρες θα μπορούσαν να επιφεληθούν από αυτή την ανάκαμψη και σε αυτήν μπορεί να βοηθήσει και ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στις ε, χώρες αυτές. Παρότι είναι χαμηλά τα έσοδα σε αυτές τις χώρες λόγω του μόχλευσης θα μπορούσαν τα ωφέλη να είναι τεράστια. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πιστικό επιχείρημα. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Πέντρο Μάρκε, Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ως Υπουργό Οικονομικών. Ευχαριστώ πολύ για την συμφωνία αυτή του Ιουλίου. Εσείς παίξατε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν, στην κινητοποίηση δηλαδή αυτή που είναι κοινή η κινητοποίηση των πόρων από τις κεφαλαγορές. Κύριε Υπουργέ, ακόμα και σε αυτά τα πλαίσια γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι η δημοσιονομική πολιτική, οι προπολογισμοί των χωρών μελών θα εξακολουθούν να πιέζονται Εξαιτία αυτής της τεράστιας κρίσης. Ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα σημαντικός, ε, κυρίως ως πρώτη αντίδραση σε αυτή την κρίση. Μόνο έτσι μπορέσαμε να διατηρήσουμε τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και του χρέους. Η πίεση όμως θα συνεχιστεί παρά τη συμφωνία αυτή, την ιστορική σημασία συμφωνία και θα συνεχιστεί και πίεση στου εθνικού προπολογισμού. Πώ βλέπετε εσεί τα δημοσιονομικά των χωρών μελών τα επόμενα χρόνια και ποιοι είναι οι δημοσιονομικοί κανόνε τη Ευρώπη που θα επιβληθούν. Ποιο είναι ο ρόλο τη νομισματική πολιτική, δηλαδή τα επόμενα χρόνια. Θα είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσουμε τη σταθερότητα αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε επίπεδο διαφόρων περιφερειών ανά την Ευρώπη. Εσείς πώς βλέπετε την νομισματική πολιτική λοιπόν. Δεν θα είναι πια νομι... παραδοσιακή όπως την ξέραμε, γιατί τώρα έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νομίζω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα από την νομισματική πολιτική, συγγνώμη, τη δημοσιονομική πολιτική στην Ευρώπη. για την πολιτική της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας θα ήθελα να μην εκφραστώ, διότι είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά θα έλεγα ότι η εντολή της ΕΚΤ ε, βασίζεται στις συνθήκες ε, όπου και έχει παγιωθεί. Τώρα όσον αφορά το ερώτημα του πώς μπορούμε να εμποδίσουμε να βρεθούμε σε δύσκολη κατάσταση για τα κράτη-μέλη, επανέρχομαι στην απόφαση που ελήφθη φέτος. Είπαμε ότι θέλουμε και grants 390 ε, δισεκατομμύρια ευρώ ως κομμάτι της συνολικής προσφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη-μέλη ώστε να ε, αποφευθεί να είναι αυτή η δωρεά υπερβολικά μεγάλη. Τώρα βρισκόμαστε εν μέσω της κρίσης και θεωρώ ότι είναι μια στρατηγική που μπορούμε να υπερασπιστούμε. Ε, ήταν ρεαλιστική η αντιμετώπιση μας και χρησιμοποίησαμε τις ευελιξίες που μας προσφέρει η Ευρώπη όσον αφορά το θέμα της σταθερότητας. Το ίδιο θα κάνουμε σίγουρα και του χρόνου και μετά θα δούμε. Thank you very much. Now, Nick Wallace from GUE. Ευχαριστώ πολύ ο Nick Wallace από την GUE. Thanks very much, President, and thanks, Mr. Schultz, uh, for your presentation so far. Um, with the COVID-19 pandemic that still grips Europe, Uh, COVID-19 πού θα οδηγήσει. Η κρίση θα γίνει πιο σοβαρή από ό,τι είναι τώρα. Απαιτεί ριζοσπαστικές αλλαγές και απαντήσεις από όλα τα θεσμικά όργανα. Να αποφύγουμε τη λιτότητα, τις ε, νεοφιλελεύθερες πολιτικές που οδήγησαν και στις προηγούμενες κρίσεις οι Υπουργοί Οικονομικών ε, της Γερμανίας θα πρέπει να αλλάξουν τακτική τώρα. Η κοινωνική συνοχή στις χώρες μέλη είναι ζωτική σημασίας. Ο συνασπισμός ζήτησε να αποφύγει παραπάνω νόμους και δυσκολίες στους εργαζόμενους η Γερμανική Προεδρία θα βοηθήσει να αποφευθούν οι κανόνες λιτότητας αυτή τη φορά. Αυτό που κάνουμε αυτή την περίοδο είναι ακριβώς μια ιδιαίτερα επεκτατική, αν θέλετε, πολιτική σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση κρίσεων. Ε, δηλαδή, ότι προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε κονδύλια σε ευκολότερε περιόδου, έτσι ώστε ακριβώ σε τέτοιε περιόδου κρίσεων να έχουμε τέτοιου είδου κονδύλια στη διάθεσή μα. Ε, και νομίζω πω ε, ε, πολύ γρήγορα, όταν ξεκίνησε η κρίση, καταλήξαμε στο συμπεράσμα ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να κινηθούμε. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και φέτο και του χρόνου. Να έχουμε δηλαδή μια κοινή αντιμετώπιση τη κρίση και να δημιουργήσουμε τι απαραίτητε προποθέσει για την ανάκαμψη τη Ευρώπη. Και επιτρέψτε μου να συμπληρώσω κάτι ακόμα. Όσο περισσότερο κάνουμε κάποια πράγματα από κοινού, τότε ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να ε, διευκρινίζονται και κάποια άλλα ζητήματα, όπω για παράδειγμα αυτό το θέμα τη ελάχιστη φορολογία των επιχειρήσεων. Είναι κάτι το οποίο θα διευκρινιστεί έτσι ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον να συνεργαστούμε και ακόμα πιο στενά μεταξύ μα. Ευχαριστώ. Now our last request, Monica. Τελευταία, Μερικά εδώ, Renew. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Σόλτς που είστε εδώ σήμερα. Η ερώτησή μου αφορά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η πανδημία έδειξε τα προβλήματα που είναι διασυνοριακά. Εγώ είμαι από το Λουξεμβούργο και έρχονται εκεί 200.000 άνθρωποι να δουλέψουν από τη Γαλλία, τη Βελγία και τη Γερμανία καθημερινά και Λόγω του lockdown, πολλοί άνθρωποι χρειάστηκαν να δουλέψουν με τηλεεργασία. Πολύ περισσότεροι από ό,τι έδειξαν οι αριθμοί μέχρι σήμερα. Από όσο προβλεπόταν. Με αυτούς τους αριθμούς αλλάζουν ε, το καθεστώς φορολόγησής τους και ασφάλειας και δεν είναι υπέρ τους μέσω συγκεκριμένων συμφωνιών με τις γειτονικές χώρες ε, αποφεύχθηκε ε, να τιμωρηθούν οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Σόλτσο, αυτή η αβεβαιότητα, το μη αναγκαίο στρες ε, για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες μας πρέπει να αποφευχθούν στο μέλλον. Ε, αυτός ο δυσυνοριακός συντονισμός πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η διασυνορική συνεργασία. Δεν βλέπετε ότι υπάρχει ανάγκη για μια μόνιμη λύση στην Ευρώπη. Το δικαίωμα του να υπάρχει τουλάχιστον μία ημέρα τηλεργασίας για όλους χωρίς να τιμωρούνται σε θέματα ασφάλειας ή κοινωνικού ε, καθεστώτος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και φορολογικού καθεστώτος. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, προσπαθούμε να βρούμε, έχουμε βρει ρεαλιστικές λύσεις για τη σημερινή κατάσταση. Κάτι που βοήθησε πολλούς ε, ε πολίτες και πολλά κράτη-μέλη και χαίρομαι που αυτό έγινε πάρα πολύ γρήγορα σχετικά. Τώρα το θέμα του τι θα γίνει στο μέλλον Κατά πώς θα υπάρξει ένας γενικός κανονισμός. Δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό. Ειλικρινά, οι φορολογικοί κανόνες είναι τόσο διαφορετικοί σε κάθε χώρα που δεν είναι τόσο απλό να υπάρξει ένα μέτρο για όλες τις διασυνοριακές περιπτώσεις. Η τηλεργασία είναι σημαντική. και θεωρώ ότι η πρόταση πρέπει να συζητηθεί. Δεν έχω συγκεκριμένη άποψη. Φυσικά έχουμε τους σημερινούς κανόνες ε, όπου πρέπει να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων που χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα της διασυνορικής εργασίας στην Ευρώπη. Ωστόσο υπάρχει και κάποια διατησία που πρέπει να αποφευχθεί με αυτό και έτσι τα πράγματα είναι λίγο ακόμα περίπλοκα. Chair, Πρόεδρος, Συγγνώμη, μερικές φορές η σύνδεση μου κόβεται. Είναι αδύναμη, λέει η Πρόεδρος. Ωραία, ολοκληρώσαμε λοιπόν τον γύρο αυτό ερωτήσεων και απαντήσεων. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Σόλτς για το ότι ήταν διαθέσιμος να είναι μαζί μας σήμερα και τους ευρωβουλευτές για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις τους και τη συζήτηση. Κύριε Σόλτς, όπως διαπιστώσατε κι εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μαζί σας όταν μιλάτε για αύξηση της ολοκλήρωσης ή περισσότερη αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι μάχες που δίνουμε κι εμείς εδώ, οπότε θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί ξέρουμε ότι εκεί βασίζεται το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται αλληλεγγύη και όχι μόνο, πολύ περισσότερα. Έχει να κάνει με την εσωτερική αγορά, την νομισματική ένωση κλπ. κλπ. Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε ότι οι οικονομίες μας είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Και όταν παίρνουμε μέτρα για να προστατεύσουμε την εσωτερική αγορά, είναι κάτι προς όφελος όλων. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεργαστούμε και θα βρεθούμε ξανά και ξανά τους επόμενους μένες. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να κηρύξουμε την λήξη της συνεδρίασης.